Bene. Ωραία, λέει ο ε, Πέστεψε ο κύριο Επίτροπο, είμαστε όλοι εδώ, οπότε έχουμε τώρα την τρίτη συζήτηση για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοκρατίας και κρατου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 135 του κανονισμού. Σύμφωνα με την ε, μεσιάταξη θα συζητήσουμε για την ε, Μαλαισία. Θα μιλήσουν πρώτα-πρώτα οι συντάκτες της πρώτης ψηφίσματος. Κορά. Ευχαριστώ Προέδρο. Οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής